γίνει αύριο. Το επόμενο είναι η έκθεση Κάσμαν για την ε, επίτευξη των εμψηφιακών στόχων τη χιλιετία ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο τη προετοιμασία για τη συνάντηση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του 2010. Το λόγο έχει ο συγητή Μάικλ Κάσμαν για τέσσερα λεπτά. Thank you, Madam President. Um, can I say, as I begin, I think we should really call these not millennium, millennium development. Θα ήθελα να πω καταρχήν πρόεδρε ότι δεν πρέπει να μιλάμε για στόχους της χιλιετίας αλλά για προκλήσεις ε, της χιλιετίας. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, στην ουσία επανεξετάζουμε γιατί πρόκειται το 2000 όταν ε, γνωρίζαμε μία οικονομική ανάκαμψη, κάναμε, προβήκαμε μάλλον σε δεσμεύσεις. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Είμαστε πέντε χρόνια πριν από την προθεσμία, το 2015, όταν μιλήσαμε για αυτές τις βασικές προκλήσεις. Μιλάμε για την ακραία φτώχεια και την ε, πείνα. Ε, πρόσβαση στην πρωτοβάθμια ε, εκπαίδευση, αντιμετώπιση της παιδικής θνησιμότητας, αντιμετώπιση του AIDS, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και εταιρικές σχέσεις. Και μιλάμε και για φιλοδοξίες της χιλιετίες που παραμένουν φιλοδοξίες και όχι στόχοι. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη βδομάδα θα ορίσει μία ενία στάση ε, εν ώψη της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο. Όμως ε, δεν υπάρχει επαρκής ε, ε, δέσμευση σε σχέση με το 0,7% του ΑΕΠ που είχαμε αναλάβει για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βρισκόμαστε πολύ κάτω από το στόχο αυτό στη μέση της πορείας μας. Έχει επιτελεστεί κάποια πρόοδος, όμως οι επενδύσεις μας, και το λέω αυτό με πλήρη σύνεση, έχει αποδώσει, ιδιαίτερα ως προς τη μητρική υγεία. Έχουμε αντιμετωπίσει την παιδική θνησιμότητα. Οι δείκτες είναι χαμηλοί, αλλά επιτέλους μειώνεται ο αριθμός της παιδικής θνησιμότητας. Δεν χρειαζόμαστε όμως περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, δεσμεύσεις, αλλά και επιπρόσθετη χρηματοδότηση που σχετίζεται με την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και αυτό ε, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε όχι τι κάναμε μέχρι τώρα, αλλά ποιος δρόμος, πόσος δρόμος υπολείπεται. Θα πρέπει να δούμε και τα θεσμικά μας προβλήματα. Μιλάμε για πολιτικές από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ε, πολιτικές οι οποίες στην ουσία είναι αντιφατικές. Δείτε τι γίνεται με την κοινή αλληλευτική πολιτική, την ΚΑΠ, τις επενδύσεις γενικότερα. Εάν δεν έχουμε συνοχή, δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Μιλάμε για επενδύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτά τα προβλήματα, από αυτή τη μάστιγα δηλαδή να μην χάνονται ζωές ανά τον κόσμο. Θα ήθελα να κατέχουμε πραγματικά, πραγματικά ηγετική, θέση, όχι έναν ελάχιστο παρονομαστή, αλλά ένα 0,7% των εθνικών ΑΕΠ, έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουμε επιπροσθέτως και να μην ορίσουμε εκ νέου την ε, την ε, πολιτική μας ως προς τις ως προς τη διπυρωτική βοήθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις μη κυβερνητικέ ανά την Ευρώπη που με υποστήριξαν. Θα ήθελα κατά την αυριανή ψηφοφορία να βάλουμε στην άκρη τις πολιτικές μας διαφορές. Δεν είναι τέλεια η έκθεση. Τίποτα το οποίο παράγουμε δεν είναι τέλειο. Απέχει πολύ από την τελειότητα. Αλλά ας μην χρησιμοποιήσουμε τις κομματικές μας διαφορές για να μην αδράξουμε αυτή την ευκαιρία να έχουμε ενιαία θέση στα Ηνωμένα Έθνη και να φτάσουμε στους στόχους ως προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες το 2015. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Κτώμα της Επιτροπής, ο Επίτροπος Πίβαλξ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Σώματος. Η σημασία ε, που έχουμε είναι ότι μπορούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε κοινού στόχου. Αυτό για τις ε, μη αναπτυγμένες ε, για τους στόχους της χειρετίας. Η γενική πρόοδος ήταν άνηση μεταξύ των διαφόρων στόχων, μεταξύ των διαφόρων περιοχών και όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2010 είναι ορόσημο. Χρειάζεται να δούμε τι πήγε καλά και τι όχι. Πού είχαμε επιτυχία και πού αποτυχία από τότε που υπεγράφει η Συμφωνία της Χιλετίας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη φάση. Πώς θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε την πρόοδο των που υστερούν αυτή τη στιγμή. Είναι επίσης σημαντικό μια πρόοδος για την επίτευξη των στόχων αυτών να διατηρηθεί. Να ενδυναμώσουμε τα διάφορα θεσμικά μέσα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης σημαντικό θα είναι η αποφυγή, η μείωση των σοκ και η προώθηση ευρείας οικονομικής ανάπτυξης. Η θαυμάσια έκθεση του κυρίου Κάσμαν ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και δίνει σημαντικέ γραμμές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προετοιμασία τη συνάντηση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο και πέραν αυτής. Χρειάζεται έντονη σύγκληση μεταξύ της έκθεσης του κυρίου Κάσμαν και της ανακοίνωσης της Εκτελεστικής Επιτροπής που έχει ήδη υποβληθεί. Χρειαζόμαστε να σεβαστούμε την ε, δέσμευση που έχουμε λάβει του 0,7% του ΑΕΠ για ενίσχυση μέχρι το 2015. Θα πρέπει η αποτελεσματικότητα της, της ε, βοήθειας να είναι μια πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε να έχουμε μια διάσκεψη για ανάπτυξη που να κατευθύνει τις ε, λήψεις αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε εκείνες τις χώρες που είναι πιο πολύ απομακρυσμένες, ιδίως εκείνες που είναι πιο ευάλωτες. Θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε εκείνους τους στόχους που δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί καθόλου. <clears throat> Συμφωνώ ότι η διακυβέρνηση είναι σημαντική για την επιτυχία και την εφορία των, της επίτευξης των στόχων της χιλιετίας. Η δυνατότητα και η δέσμευση να διακυβερνούμε αποτελεσματικά είναι σημαντική προϋπόθεση για οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια μιας ε, ε, ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη συγκεκριμένων χωρών προωθώντας την ανάπτυξη και τις επενδύσεις της χώρας στην παιδεία στην βελτίωση της υποδομής και στην προώθηση των καθαρών πηγών ενέργειας. Η δική μας βοήθεια θα πρέπει να παίξει το ρόλο καταλήτη για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τους στόχους αυτούς της χαιρετίας. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και να σας πω ότι είμαι γενικά ικανοποιημένος με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Υπάρχει σαφής δέσμευση να επιτευχθεί ο στόχος του 0,7% του ΕΕΠ μέχρι το 2015. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012 2015 όσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων. Επίσης, ένα νέο πρόγραμμα διεράσης για την επιτύχηση των επιζερκών στόχων αντιμακοτοπλίζεται στην πρόταση της Κομισιόν. Το Συμβούλιο προτίθεται να πραγματοποιήσει πραγματική πρόοδο ακολουθώντας τις ιδέες αυτές της Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας, αλλά θα πρέπει με τη δέσμη που προτείνεται να ηγηθούμε με το παράδειγμά μας στην Νέα Υόρκη και πέραν αυτής. Δεν είναι τέλεια η πρόταση αυτή, αποτελεί όμως μια βάση για πρόοδο και για άλλη μια φορά θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για την έκθεσή του αυτή για τους νομιστικούς στόχους και λιτίες. Πρώτα σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα ακολουθήσουν οι ομιλητές εκ των πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Φέντσον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσμαν για την εξαιρετική αυτή συνεργασία ως προς αυτό το θέμα. Άκρος ενδιαφέρουσα αυτή η εργασία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή λύση, αλλά είναι απόλυτα σαφές ότι υπάρχουν αποκλήσεις και διχογνωμίες. Ο κύριος Κάσμαν είπε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι, θα πρέπει να έχουμε περισσότερους. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για περαιτέρω φορολόγηση, πιστεύω κύριε Κάσμαν. Θα πρέπει οι επιχειρηματίες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Εσείς μιλάτε για ένα μορατόριουμ. Είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα σας καταρχήν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 27. Στην παράγραφο 27 λέμε ότι θα πρέπει να μην γίνονται διακρίσεις ανά ομάδες χωρών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο σε αυτές τις ε, συζητήσεις. Μιλάμε για 0,7%. Ε, εντάξει ως προς αυτό το ποσοστό, αλλά θα προτιμούσα να μιλάμε για 1% του ΑΕΠ, διότι οι πλούσιες χώρες είναι ε, κατά κύριο λόγο υπεύθυνε. και νομίζω ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να λάβουμε μια απόφαση βεβιασμένα. Έχουμε το περιθώριο μπροστά μας μέχρι το 2015. Θα πρέπει αυτή η πρόταση να είναι ένα εφαλτήριο προς τις χώρες και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για θέματα δεοντολογίας και ήθους. Οι άνθρωποι πεθαίνουν, λιμοκτονούν κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο να βιώνουμε ως μέλη του Κοινοβουλίου. Η κυρία Κρέτσου έχει το λόγο. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών για ένα λεπτό, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, ήδη ελέγχθη, η χρηματοπιστωτική κρίση που διανύουμε επηρεάζει κατά πολύ τις δεσμεύσεις των κρατών μελών ως προς την αντιμετώπιση των στόχων της χιλιετίας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ρεαλιστές μέσα στα πλαίσια και της έκθεσης. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι 10 χρόνια μετά μετά το 2000 έχει επιτελεστεί κάποια πρόοδος για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια αλλά η πρόοδος αυτή δεν επαρκεί. Αναγνωρίζουμε τα ε, αδύναμα σημεία της έκθεσης. Βλέπουμε όμως ότι η έκθεση μας δίνει εναλλακτικές για να μην δαπανούμε, λανθασμένα τους πόρους, αλλά μέσα στα πλαίσια, να τους δαπανούμε μέσα στα πλαίσια των μηχανισμών της αγοράς. Τουλάχιστον λοιπόν το ίμιση της βοηθείας θα πρέπει να αποστέλλεται στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έτσι ώστε να λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση αυτές τις χώρες ε, ως προς τα άτομα με αναπηρία, τις γυναίκες και τα παιδιά για να αποτιμήσουμε τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Σε πολλές περιφέρειες είναι κρίσιμη η κατάσταση αυτών των ομάδων. Αυτό, ε, αυτό φαντάζομαι θα λεχθεί και στα Ηνωμένα Έθνη το Σεπτέμβριο του 2006 όταν θα μιλήσουμε για θέματα ανάπτυξης και η έκθεση Κάσμαν είναι πολύ καλά διαρθρωμένη ως προς στόχους της χιλιατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ντόνσκης για την ομάδα των φιλελευθέρων για δυόμιση λεπτά. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Κάσμαν, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, οι παρατηρήσεις που θα κάνω είναι κάποιες παρατηρήσεις που συμπληρώνουν την πολύ καλή έξεση του κυρίου έξεση δεν είναι επικριτικές είναι όμως πολύ σημαντικό να έχουμε καινούριε προοπτικέ ε, προοπτικές ε, τώρα που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και όχι να παραμείνουμε σε αυτές του 20ου αιώνα γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε μια πιο εξισορροπημένη προσέγγιση στους στόχους αυτούς της χιλιετίας γιατί πραγματικά η φτώχεια πάει χέρι-χέρι με πάρα πολλά άλλα πράγματα την, ε, ε, όμως ε, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις ε, βία σε ορισμένα κράτη-μέλη, ε, βίες διαμάχες όπως είδαμε στο Κυργιστάν ε, και αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Δε, αν πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς ασφάλεια, νομίζω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος. Και όταν μιλάμε για τη φτώχεια, δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τη φτώχεια από τέτοιου είδους θεωρήσεις. Δείτε την κατάσταση στην Αλβανία και αλλού. Δείτε και άλλα πράγματα στη Μολδαβία λόγω χάρη ή στην Ουκρανία έχουμε φοβερά κρούσματα φυματίωσης Α, αυτά όλα πάνε παρέα και αν οι στόχοι της χιλιετίας δεν μας οδηγήσουν σε σταθερές κοινωνίες και σταθερά κράτη, ασφαλή κράτη, τότε δεν κάναμε τίποτε. Δεν νομίζω ότι επίσης θα πρέπει να μην λάβουμε υπόψη μας νέες προκλήσεις που αναφύονται και πιστεύω ότι ε, επίσης θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για να εξουσιοδοτήσουμε φτωχές χώρες που θα αναλάβουν από μόνες τους ευθύνες για τον εαυτό τους. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Πίμπαλξ που είστε υπεύθυνο για την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα να ήταν εδώ και ο κύριο Χόιτ, ο οποίο είναι υπεύθυνο. De που είναι υπεύθυνο για το εμπόριο, αλλά δεν πειράζει, καλωσορίσουμε και εσά. Πραγματικά δώσ, αναλάβαμε κάποιες δεσμεύσεις και δώσαμε υποσχέσεις όταν μιλούσαμε για τους στόχους της χιλιετίας. Είπαμε ότι θα εξαλείψουμε τη φτώχεια. Θα αφήσουμε τη φτώχεια στο παρελθόν. Όμως δεν φαίνεται να τα καταφέρνουμε αμέσως. Ε, ακόμη κυρίες και κύριοι μιλήσαμε, ακούσαμε τα σχόλια για το 0,7% μπορούμε βεβαίως να αυξήσουμε το ποσοστό ή να φανταστούμε καινούριε μεθόδους χρηματοδότησης αλλά όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες γι' αυτό λέω ότι εκείνο που, προ, που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να ε, φανταστούμε εναλλακτικέ μορφές συμβίωσης το fair trade παραδείγματος χάρη ή άλλου είδους ε, εμπορικές συναλλαγές ε, ε, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες για να μην χρειάζονται χρήματα από μας για να επιβιώσουν οι χώρες αυτές δεν θέλουμε να ε, ε, νομίζω ότι αν υπήρχε ένας, αν επιμέναμε σε άλλες μορφές εμπορίου θα ήταν ε, καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι αν είχαμε καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δεν δέχαμε τα τεράστια χρέη που έχουμε αυτή τη στιγμή σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Σε, βρισκόμαστε ήδη στο 2010. Μέχρι έχουμε πέντε χρόνια ακόμη. Θέλουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε μέχρι το 2015. Θα ήθελα να πω για αυτούς που βρίσκονται στην... Ε, θεωρία ότι δεν ήθιστε να ε, χειροκροτούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπάση περιπτώσει. Επόμενο επόμενος μιλητής, ο κύριος Τεβά. Ναι, κύριε Πρόεδρε, η, ο εισηγητής έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και μας... Ε, και υποστηρίζει Νομίζω ότι μπορεί να βοηθηθεί με αυτή την έκθεση του Κοινοβουλίου εν ώψη τη συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη. Συμφωνούμε πολύ με τον κύριο Κάσμαν. Μιλούμε για στόχους της χιλιετίας. Τι είναι ουσιαστική η στόχη αυτή τελικά. Εγώ νομίζω ότι αν είχαμε θέσει περισσότερους στόχους και προσπαθούσα να, επιδιώ... επιτύχουμε περισσότερους στόχους θα είχαμε καταφέρει και περισσότερα αν δείτε σε ορισμένες χώρες τα προβλήματα που υπάρχουν στους φτωχογειτονιές στην ανάγκη που έχουν οι οικογένειες να έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, το δικό τους σπίτι, οι μικρές επιχειρήσεις, τη βοήθεια που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Φαντάζομαι τα έχετε δει και εσείς τα ταξίδια σας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι φτωχογειτονιές, αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά δεν καταγράφονται και δεν αναγνωρίζονται πουθενά. Αν, αν... Ε, αν είχαμε καταγράψει όλους αυτούς τότε δεν μιλούσαμε για 8 εκατομμύρια που συζητούμε τώρα αλλά για 9 τρεις που χρειάζεται για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους. Μιλάμε για με τεράστια ποσά, ε, παραπάνω από το σύνολο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του Τόκιο κτλ. Μιλάμε εδώ για προβλήματα που ουσιαστικά βρίσκονται στο όριο έξω από το σύστημα, από το κατεστημένο, σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλο κομμάτι του κόσμου που πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ η κυρία Τσίμερ, εξονόμητος τη ομάδα της ΚΟΕ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσμαν για την υποβολή της έκθεσης αυτής ε, που εγκρίναμε στην Επιτροπή Ανάπτυξη με μεγάλη πλειοψηφία και θα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και ω Κοινοβούλιο από κοινού πριν από τη διάσκεψη αυτή στην, στον ΟΗΕ να τονίσουμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους ε, ανεπτυγικούς στόχους της χιλιετίας και να πούμε ότι ε, δεν πρέπει να ξεχνάνε τις ε, υποχρεώσει που έχουν ήδη αναλάβει, δηλαδή να συμμετάσχουν οικονομικά, να πληρώσουν το ποσοστό για να τη βοήθεια που είχαν προβλέψει. Ο κ. Κάσμαν είπε ότι βρισκόμαστε στο μείον δις αυτή τη στιγμή ευρώ. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα τι θέλουμε. Θέλουμε Αυτή οι αναπτυξιακοί στόχοι να επιτευχθούν μέχρι το 2015. Δεν θα επιτρέψουμε να βληθεί ο στόχος αυτός λέγοντας ότι υπάρχει κρίση και γι' αυτό εμείς ως εθνικές ε, κυβερνήσεις δεν είμαστε σε θέση να πετύχουμε αυτό που θέλουμε ή και ότι ε, έχουμε το δικαίωμα να αναβάλουμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ε, ζουν σε φτώχεια, πεινάνε και σε ορισμένες περιοχές του κόσμου όπως νότια της Σαχάρας αυξήθηκε η ένδια τα περισμένα χρόνια αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πραγματικά να ζητήσουμε επιμόνως αυτό που έχουμε ορίσει και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους δύο από τις αντιληστικές ομάδες να μην ε, επιβάλλουν τις τροπολογίες τους που αποδυναμώνουν την έκθεση αυτή γιατί η έκθεση νομίζω αποτελεί μια ισορροπημένη ε, λύση μεταξύ των απαιτήσεων, της πίεσης που θέλουμε να ασκήσουμε και δεν πρέπει να αφαιρέσουμε τίποτα. Εγώ θα πήγαινα και πολύ πιο μακριά σε ορισμένα σημεία θα ήθελα να ζητήσω συγκεκριμένα ότι δεν θα πρέπει να υπογράφουμε καμία άλλη συνθήκη η οποία να μην εξυπηρετεί την επιβολή των στόχων ανάπτυξης χιλιτίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεπή πολιτική, όχι μέσα στα πλαίσια ενεψιακής ε, πολιτικής μόνο, αλλά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θέλουμε να καταπονεμήσουμε την υποανάπτυξη και την ένδυα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπατέν για την Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας για 1,5 λεπτό. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τους αναπτυξιακούς στόχους ε, όπως ορίστηκαν το 2000, αλλά πιστεύω ότι οι στόχοι αυτοί δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέχρι το 2015. Αυτό είναι ανέφικτο. Πέρα από, το μη, από τη μη ρεαλιστική προθεσμία υπάρχει και το θέμα των χρημάτων που θα πρέπει να δαπανηθούν. Από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα. Οι περισσότερες χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού και της ε, πτώχευσης και μόνο αν γίνουν περικοπές θα αναστραφεί η κατάσταση. Άρα ε, τι κάνουμε, περιμένουμε από τις πιο φτωχές χώρες να γίνουν πιο ευήμερες και να τονώσουν την παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πρέπει να φορολογήσουμε τις επιχειρήσεις που είναι επικερδείς και να τις διώξουμε εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας. Θα πρέπει όμως να μειώσουμε τα προστατευτικά μέτρα και να περιορίσουμε το εμπόριο με τις φτωχότερες χώρες. Θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία που πραγματικά στραγγαλίζει τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στην Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, και η Ιταλία να επανέλθουν στον κόσμο της ε, οικονομική πραγματικότητα και βεβαίω το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν. Πάμε στους ε, επόμενου ομιλητέ. Ο κύριο Φίσας έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της φτώχειας και οι άλλοι στόχοι της ε, χιλιετίας θα πρέπει να μας ενώσουν όλους και λυπάμαι, διότι ορισμένες πολιτικές ομάδες εισήγαγαν θέματα τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ομοφωνή, όπως το θέμα των αμβλώσεων για να ελέγξουμε την γεννητικότητα ή την φορολόγηση ως προς τις συναλλαγές και τα μερίσματα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό και δεν είναι και εύκολα εισπράξιμο. Εάν λοιπόν θέλουμε να ελέγξουμε την κατάσταση, ιδιαίτερα ως προς τα μεγάλα χρηματοοικονομικά μπλοκ, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις χώρες που μπορούν να εφαρμόσουν όλα αυτά τα θετικά σημεία. Είναι κρίμα να μην φτάσουμε σε μια ομοφωνία, σε μια τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σασόλη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο καθώς και τον εισηγητή Κάσμαν διότι μας μίλησε για τη σημασία της διάσκεψης κορυφής της Νέας Υόρκης η Ευρώπη έχει μια μεγάλη ευκαιρία να φανεί ως ενιαίος και μοναδικός εταίρος σε αναπτυξιακά θέματα. Μιλάμε για ένα δις ανθρώπων που πλήττονται από χρόνια λιμοκτονία και θα πρέπει να δούμε τώρα και να αποτιμήσουμε και την αρνητική, τον αρνητικό αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι στόχοι του 2000 ήταν φιλόδοξοι σίγουρα, αλλά μόνο οι χώρες δωρητές θα μπορούσαν να τηρήσουν αυτούς τους όρους. Υπό το φως αυτών των δεδομένων, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται μακριά από τους στόχους. Λυπάμαι που η χώρα μου, η Ιταλία, βρίσκεται σε ένα 0,16% του ΑΕΠ θα πρέπει να δεσμευτούν όλες οι αναπτυγμένες χώρες. Να φτάσουμε στο 0,70% του ΑΕΠ μέχρι το 2015 όπως όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλες οι χώρες έχουν ηθικό χρέος προς κάτι τέτοιο έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη δέσμευση που αναλάβαμε το 2000 και να προωθήσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια γενικότερα. Η κυρία Κέλλερ για 1,5 λεπτό. Η αναπτυξιακή στόχη της χιλιατίας δεν είναι τέλειοι, αλλά μπορούν να προσμετρηθούν και να αποτιμηθούν. Άρα βλέπουμε ότι δεν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Τα θεσμικά όργανα αλλά και εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες προς αυτούς τους στόχους, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση του τομέα της αλίας, να βοηθήσουμε τους άνδρες και γυναίκες ε, αλίης σε όλες τις χώρες. Επίσης, την ΚΑΠ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη βιώσιμη γεωργία για να απομακρύνουμε τις άμεσες και έμεσες επιδοτήσεις. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μεταφορά τεχνολογίας και ιατρικής περίθαλψης. Δεν υπάρχει μητρική υγεία χωρίς δικαιώματα των γυναικών. Όλα αυτά δείχνουν ότι η αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι ένας μικρός τομέας μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την πολιτική σε όλες μας τις κοινοβουλευτικές επιτροπές χωρίς ε, συνοχή, πολιτική συνοχή όπως ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν θα φτάσουμε πουθενά. Και αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να ξέρω από την Επιτροπή τι δράσεις θα αναλάβει μετά το 2015. Ο κύριος Γουαρό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι λυπηρό να συνειδητοποιούμε ότι στα δύο τρίτα του δρόμου χρονικά είμαστε τόσο μακριά από τους τελικούς στόχους παρόλο που είμαστε σε περίοδο κρίσης τουλάχιστον εκείνο που θα έπρεπε να, είχαμε, να, να, να επιμείνουμε να γίνει είναι η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των φτωχών χωρών να τηρηθούν το 0,7%. Από την άλλη μεριά για την εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ ε, εγώ θα έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος των κονδυλίων με, στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών ε, αφιερώνεται ουσιαστικά στο εμπόριο ενώ θα έπρεπε να αφιερώνεται σε αναπτυξιακέ δράσεις και εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λιγάκι την ισορροπία εκεί Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος ο κύριος Πρέντα για δύο λεπτά ο επόμενος ομιλητής Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό στην η συνεδρίαση της Νέας Υόρκης η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ενιαία θέση και να πούμε ότι ε, θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας έναν των αναπτυσσομένων χωρών. Η απόφαση του Συμβουλίου που πάρθηκε σήμερα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε η Ευρωπαϊ... Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρας, εταίρος συγγνώμη, Δεν μπορεί να θετήσει τις υποσχέσεις τους. Θα, και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε και τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε, για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές. Α, την άλλη μεριά πιστεύω ότι θα πρέπει η διάσταση προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ε, είναι κομμάτι όλων των δράσεών μας, όλων των προγραμμάτων μας. Θα πρέπει να, προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, παντού και να βοηθήσουμε τους φτωχούς αυτού του κόσμου να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια αλλά υπάρχουν και ορισμένα άλλα πράγματα που θα πρέπει να προσέξουμε στο κομμάτι 8 της παραγράφου 9 αυτό που αναφέρεται δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε επίσης στην παραγράφο 9 δεν αναφέρεται κάτι που δεν το υποστηρίζουμε απολύτως γιατί οι χώρες αυτές θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και να αντιμετωπίσουν μόλες τους τα, τις προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νόιζερ για ένα λεπτό τώρα. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, η επίτευξη των ε, στόχων του, της χιλιετίας σαφώς εξαρτάται από το πόσο χρήμα, τι ποσά θα δώσουν οι βιομηχανοποιημένες χώρες για την αντιμετώπιση προβλημάτων είτε ασθένειες είναι αυτές είτε οτιδήποτε άλλο. Όμως φοβάμαι ότι κάποια πράγματα δεν θα μπορέσουν να γίνουν. 50 δις δολάρια, αμερικανικά δολάρια τάξαμε στις, στις ε, ε, αναπτυσσόμενες χώρες για φέτο. Μόνο 36 θα μπορέσουν να δοθούν. Οι πλούσιες χώρες λένε ότι διαθέσουν 0,7% για τις φτωχότερες χώρες. Δεν θα γίνει ούτε αυτό και υπάρχουν δυστυχώς κακά παραδείγματα όπως είναι η χώρα μου, ε, όπως είναι στη χώρα μου. Η, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία μπορεί να δουλεύει καλύτερα, ίσως πρέπει να τους μιμηθούμε. Γεραίρο. Κύριε Κάσμεν, κύριε Πρόεδρε, το 2000 ορίσαμε τους στόχους που θα έπρεπε να επιτύχουμε για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια, τον αποκλεισμό και την ανισότητα. Όμως αναλάβαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις χωρίς να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Δημιουργήσαμε όμως μία δυναμική που αγκάλιασαν κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές και ίδιες οι αναπτυσσόμενες χώρες. Προχωρήσαμε, αλλά όχι επαρκώς και η κρίση μας κάνει να παλινοδίσουμε. Ακούσαμε τους ευρωσκεπτικιστές και πολλούς εγωιστές που μας είπαν ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ρεαλισμός σήμερα σημαίνει να αλλάξουμε την χειροπιαστή πραγματικότητα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε αύριο με την ψήφο μας αυτή την έκθεση. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το Συμβουλίο διότι το 2015 θα πρέπει να επιτύχουμε αυτό που είχαμε πρόθεση να επιτύχουμε το 2000. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο τμήμα Κασουδιάη. Ορισμένοι έχουν ζητήσει το λόγο ήδη. Ο κ. Νικολέσκου, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ στο σημείο 22 της έκθεσης που αναφέρεται στην ε, μείωση των επιδοτήσεων των ε, αγροτικών εξαγωγών και άλλων πτυχών της αγροτικής πολιτικής. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς επιδοτήσεις αυτές, ιδίως αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί υποφέρουν από τις, ε, από τις διατάξεις που επιβάλλουν για την ποιότητα των προϊόντων και την ευμάρεια των ζώων και βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολε θέσει όσον αφορά την εξωτερικό ανταγωνισμό. Πιστεύω λοιπόν ότι αν τερματίσουν οι επιδοτήσει αυτέ θα υπάρχουν σημαντικότατε και αρνητικέ επιπτώσει στου παραγωγού και παρακαλώ να καταψηφίσουν. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρο. Κύριε Μαγκίνε, ένα λεπτό. Πρόεδρο, ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή τον Γιώργο Κάσμα για την έκθεση αυτή και την παρουσίαση της έκθεσής του. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τις παραγράφους 49 και 50. Νομίζω ότι η η τη ε, δήλωση για την επιστημιστική ασφάλεια είναι πιο σαφή από ότι τα άρθρα αυτά. Γιατί όσο πάει, δαπανούνται μικρότερο τμήμα τη αναπτυστική ε, βοήθεια εκεί που θα χρειαζόταν περισσότερο. Δηλαδή για την επιστημιστική ασφάλεια και για την ε, παραγωγή των μικρών παραγωγών. Εμείς λιμιώνουμε από 17% το 1980 σε 3% έχουμε μειώσει τον τύπο αυτό της ε, βοήθειας. Θα μας πει ίσως η Κομισιόν ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουν για να τον επιτοπίσουν ε, και βλέπω πολλούς να γράφουν καταφατικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ε, πείνα σε αγροτικές περιοχές όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι τις ανάγκες τους αν είχαν τις απαραίτητα μέσα στη, διάθεσή τους. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Αρσένης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσμαν για μια εξαιρετική δουλειά. Πρέπει πραγματικά να υποστηρίξουμε όλοι ένθερμα αυτή την έκθεση, να στείλουμε το μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να μείνουν συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους για την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Εμέσω μέσω αυτής της οικονομικής κρίσης που πρέπει να μην ξεχνάμε μπορεί να πλήττει εμά, αλλά πλήττει και τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι τα δικά τους προϊόντα που πολλές φορές δεν καταναλώνουμε είναι και σε αυτές τις χώρες που αυξάνεται η φτώχεια ε, και αυξάνονται όλες αυτές οι επιπτώσεις όλες αυτές οι δύσκολοι δείκτες που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με, τα, με τους στόχους χιλιετίας. Την ίδια στιγμή η κλιματική αλλαγή που εμείς προκαλέσαμε επιδεινώνει την πρόσβαση στη τροφή, σε νερό, στις υπηρεσίες υγείας, επιδεινώνει την ίδια την υγεία. Χρειαζόμαστε πλέον πόρους λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή να προσαρμοστούν αυτέ οι χώρε να βοηθήσουμε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά να είμαστε συνεπεί και με του στόχου χιλιετία και αυτό θα, αυτή οι πόλη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη δήλωση τη κυρία Χέντεγκαρτ, τη Επιτρόπου, ότι η Επιτροπή στηρίζει αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλβέστρος, για ένα λεπτό. Είναι πολύ ε, δύσκολο να ανταποκριθούμε. Θα πρέπει όμως όλες οι πολιτικές ε, ομάδες να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση. Αλλά σε αυτή την έκθεση υπάρχουν στοιχεία καθαρά ιδεολογικά. Το άρθρο 42 μιλά για την άμβλωση και για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Βλέπουμε όμως ότι εισάγονται αρχές τις οποίες ε, δεν συμμεριζόμαστε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη γεννητικότητα, τη μητρική υγεία και πιστεύω ότι τα κράτη θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τον οικογενειακό προγραμματισμό ε, μέσω του χαπιού Πιστεύω όμως ότι η ευγονική θα πρέπει, δεν μπορεί να υποστηρίζει το θάνατο αλλά τη ζωή. Δεν θα πρέπει να ε, ξαναγκάζουμε στην άμβλωση γυναίκες οι οποίες δεν το επιθυμούν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Παπενικολάου για ένα λεπτό. Τελικά το είπατε σωστά κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Πράγματι, κυρίε και κύριοι, η αποτυχία επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων πρέπει να μα προβληματίζει έντονα τόσο λόγω τη απροθυμία κάποιων κρατών μελών όσο και λόγω των αντικειμενικών οικονομικών αδυναμιών προκαλεί η κρίση. επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο και συγκεκριμένα στον ενδιάμεσο στόχο 8 που αναφέρεται στη βοήθεια των αναπτυγμένων χωρών προ αναπτυσσόμενες. αναπτυσσόμενε αναφέρθηκαν ήδη αρκετοί συνάδελφοι σε αυτό. αν και ο ενδιάμεσο στόχο κυρίε και κύριοι φιλοδοξούσε στην αύξηση τη βοήθεια προ αναπτυσσόμενες αναπτυσσόμενε χώρε στο 0,56% του παγκόσμιου αεπ σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο βρισκόμαστε μόνο στο μηδέν τρία δηλαδή στο μισό του προβλεπόμενου στόχου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο στο. μηδέν τέσσερα και βεβαίω σε αυτό έχουμε και το ηθικό δίλημα κατά πόσο οι πόροι που διαθέτουμε ε, αφιερώνονται εκεί που πρέπει σε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη και ε, δεν αναλώνονται άδικα μέσα από διεφθαρμένες πρακτικές και κυβερνήσεις. καταλήγω λοιπόν λέγοντας κυρία πρόεδρε χρειαζόμαστε αναπτυξιακή λογική οικονομική προσέγγιση στα δεδομένα αυτά και όχι απλώς κάποιες φορές να καλύπτουμε τις τύψεις των αναπτυγμένων χωρών προς τα αναπτυσσόμενες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όμπερμα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Οι στόχοι της χαιρετίας ε, είναι εν μέρη να δώσουν στους φτωχούς των φτωχοτέρων μια αξιοπρεπή ζωή στις χώρες τους. Ε, είναι σημαντικό αυτό. Θα ήθελα να τονίσω και την καταπολέμηση βαριών ασθενών, ιδίως στις μητέρες και στα παιδιά. Επίσης θα πρέπει να ε, εξετάσουμε την αγροτική πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, όποιο δίνει αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να περιμένει και στην εργασία. Περιμένω λοιπόν στην εργασία εκείνων που δέχονται την ε, βοήθεια αυτή με την επιστροφή παρανόμων μεταναστών στις χώρες τους. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δεν πρέπει να εξαφανίζονται κάπου χωρίς να ξέρουν ακριβώ τι γίνεται θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η οικονομική κατάσταση των κρατών μελών είναι πάρα πολύ δύσκολη και όσο πιο, πολύ εμείς, πιο γρήγορα εμείς θα αποδείξουμε, τόσο πιο γρήγορα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και εκείνους που μας χρειάζονται. Πρώτα σας ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε τώρα την συζήτηση Καρσδάη. η κυρία Κάνεμπα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα επίση ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κάσμαν. Αναψυχή βοήθεια και καταπολέμηση ένδυα δεν πρόκειται να είναι μια πολιτική ε, μια πολιτική απλώς ελεημοσύνης. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ζουν αξιοπρεπώς, να εργάζονται αξιοπρεπώς και να μπορούν να ε, ε δημιουργούν τις, ε, τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους δεν πρέπει εμείς να κατασπαλούμε τις ενέργειές μας ε, για να βρούμε δικαιολογίες γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί ή δεν θέλουμε και όλοι. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όση ενέργεια έχουμε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή για την χρηματοδότηση της ψυχικής βοήθειας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πιμπάλξ, ο Επίτροπος, για να κλείσει τη συζήτηση. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Θα αναφερθώ σε ένα-δυο σημεία μοναχά που νομίζω ότι χρήζουν διευκρινήσεων. Η στόχη αυτή θα πρέπει και μπορούν να επιτευθούν. Αυτό δεν είναι μοναχά η δική μου άποψη, είναι και η άποψη των Ηνωμένων Εθνών, είναι και η άποψη των ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, ζητήσει ζητήσει να δεσμευθεί το 0,7%. Ξέρω ότι εδώ μπαίνουμε στα χωράφια της εθνικής κυριαρχίας. Αλλά εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητήσει κάτι τέτοιο, τότε ποιος θα το ζητήσει με τόσο ισχυρή φωνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξουσίες δεν θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να υποτιμάτε τις εξουσίες σας εδώ γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μιλήσετε επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την υποσαχάριο Αφρική Ξέρω ότι υπήρξαν πολλές προσπάθειες και απογοητεύσεις, αλλά είμαι καινούριο αν θέλετε, σε αυτά τα καθήκοντα προσπάθησα να δω ποια είναι η κατάσταση κοίταξε το πικιοκρατικό παρελθόν το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην ιστορία νομίζω λοιπόν ότι η υποσαχάριος Αφρική χρήζει περισσότερης προσοχής τώρα για τα θέματα του εμπορίου και του δίκαιου εμπορίου και τα λοιπά Ξέρουμε ότι μέχρι τώρα δεν έγιναν, έγιναν κάποια πράγματα για το εμπόριο, αλλά τελικά δεν βοήθησαν και πάρα πολύ. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δίκες συνθήκες για δίκες εμπορικές συναλλαγές και να τονίσουμε την ε, περιφερειακή διάσταση του εμπορίου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί Τώρα, η φοροδιαφυγή ακούστηκε και οι παράνομες διαδρομές κάποιων χρημάτων. Νομίζω ότι και η ομάδα των 20 και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουμε να καταπολεμήσουμε την ε, φοροδιαφύγη επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν σωστά κτηματολόγια και καταγραφή της κατάστασης διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε Νομίζω ότι η υπάρχει σαφής ε, διάσταση, ε, διάσμευση πάντως ε, σχετικά με την επιστημιστική ασφάλεια που αναφέρατε και την ε, βοήθεια σε τρόφιμα και τα λοιπά. Υπάρχει δέσμευση και αυτό που θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Κάσμαν ότι κοιτάξτε να δείτε ακόμη και αν υπάρχουν μικρές διαφορές αυτό δεν θα πρέπει να διασπάσει την ενότητα του Κοινοβουλίου, την ενότητά μας γιατί αυτό θα σημάνει ότι δεν θα επιτύχουμε τέλος πάντων για όλους τον κόσμο και για τους φτωχότερους τους στόχους μας. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τα καταληκτικά σας λόγια. Ήταν άκρος ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σκιώδης, ε, την κυρία Τζίμε, Σαγκεντίνη και τους ε, άλλους. Πολλές φορές παραλείπω μερικούς. Η ηλικία φταίει γι' αυτό. Δεν θέλω να ζήσω περισσότερα χρόνια και να ζήσω μεγαλύτερη φτώχεια, μεγαλύτερη πείνα, λιμοκτονία και γυναίκες που ζουν δραματικές στιγμές. Θα ήθελα να πω σε όσους μίλησαν με κάποια επιφύλαξη για στοιχεία αυτής της έκθεσης, ας μην γυρίσουμε την πλάτη στους πολίτες μας και να τους πούμε ότι δεν τα καταφέραμε, δεν συμφωνήσαμε, διότι υπήρχαν στοιχεία της έκθεσης τα οποία δεν μπορούσαμε να προσυπογράψουμε. Τι μήνυμα αποστέλουμε προς τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, που δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, σε τροφή, σε στέγη και ούτω καθεξής. Αλλά κάπου στις Βρυξέλλες έγιναν συζητήσεις οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε συμφωνία για την πλειοψηφία του πλανήτη. Θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να λάβετε υπόψη ότι αύριο θα ήταν σκόπιμο να υπερψηφίσετε αυτή την έκθεση. Όχι για μένα, γιατί ο Μάικλ Κάσμα θα γυρίσει στο σπίτι του όπου έχει υγειονομική περίθαλψη, ε, έχει φως, έχει νερό, έχει φαΐ και εν πάση θα με περιθάλψουν όταν μεγαλώσω και είμαι ηλικιωμένο. Αλλά σκεφτείτε αυτά τα παιδιά που πεθαίνουν από ελονοσία, από, από διάρρεια, από AIDS ή τη στιγμή που γεννιούνται τη νέα γυναίκα η οποία δεν είχε πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μη σκεφτόσαστε εμάς, σκεφτείτε αυτούς εκτός αυτού του χώρου. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έχει κλείσει και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε σε δεύτερη ανάγνωση την έκθεση